Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Νομίζω είμαστε όλοι που πρέπει εδώ. Οπότε, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Βάλτε καλύτερα τα ακουστικά σας. Ε, Έχουμε σήμερα διερμηνία γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, πορτογαλικά, φιλανδικά, εστονικά και πολλά άλλα. Επίσης ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και θα ήθελα να σας πω αν είδατε τις αποφάσεις ε, των συντονιστών της 28ης 8ης Νοεμβρίου ε, ε, εφόσον δεν έχω λάβει παρατηρήσεις θα θεωρήσω ότι γκρίνονται. Ε, να σας πω επίσης ότι σας εστάλει ε, μέσω mail και ευχαριστώ τους συναδέλφους και τη γραμματεία η έκθεση στα αγγλικά για την ε, αποστολή στην κολονία ε, που έγινε 18 και 20 Μαΐου του 2016. Σας στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα. Να σας πω και κάτι ακόμα ενημερωτικά, αν και ακόμα συνεχίζεται η διαδικασία για τον προϋπολογισμό, αλλά θεωρώ πως είναι σκόπιμο να σας θυμίσω ότι προσθέθηκε στην τελευταίο τριμερή μια συμφωνία για τον προπολογισμό του 2017. Ξέρετε πόσο έχει αγωνιστεί η Επιτροπή Πολιτισμού ώστε να αυξηθεί Αναυξηθούν τα προγράμματα. Για την ώρα τα νέα που έχουμε είναι ότι μετά από την περικοπή που ανακοίνωσε για το Erasmus Plus το Συμβούλιο έχουν αποκατασταθεί 50 εκατομμύρια από αυτά που είχε κόψει το Συμβουλίο και για την πρωτοβουλία για τους νέους 5 εκατομμύρια επιπλέον σε σχέση με το ΔΙΣ που είχε προβλεφθεί για όλο το φάσμα μέχρι το 2020 και 500 ε, εκατομμύρια συγγνώμη προσθέθηκαν και μετά ε, για τις, όλες τις νέες σημαντικές πολιτικές που έχουν ξεκινήσει η, τα κονδύλια που προβλέπονται είναι πολύ χαμηλά και για την ώρα ξέρουμε ότι έχουν προσθεθεί τρία επιπλέον εκατομμύρια για το Multimedia Actions και συγκεκριμένα για το Aeronet Plus που όπως θα θυμάστε όλοι ζητήσαμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό αλλά ακόμα δεν έχουμε νέα για τα υπόλοιπά μας προγράμματα. Συνεχίζουμε λοιπόν την πίεση αφού δεν έχουν κλείσει οι διαπραγματεύσει, αν και έχει βρεθεί ένα εκατομμύριο στην πολιτιστική κληρονομιά στη γραμμή πολιτισμός. Είναι θετικό ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς πού πώς, πώς θα γίνει, αν θα είναι επιπλέον ή αν θα είναι μέσα στο σύνολο του κονδυλίου. Πάντως υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, όπως το είχαμε ζητήσει για το 2017. Αυτά είναι τα νέα που έχουμε και μετά, έπειτα έχουμε και τους συγητές μας, οι συγητές και οι σκιώδες. Ε, νομίζω πως ήταν σωστό να σας ενημερώσω η Σαμπίν. Ένα σύντομο σχόλιο για τις προφορίες αυτές. Εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και πάλι ε, ότι αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες ε, κάποιοι ένα ε, μέσω ενημέρωσης της Βρυξέλλες διαδίδει κάτι ψευδείς ειδήσει για το εράσμος. Τι έγινε, δεν λειτουργεί η διερμηνία. Ήθελα λοιπόν να πω μόνο το εξή. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί κυκλοφόρησε ένα ράδιο αρβίλα ε, και έχει αναστατωθεί ο κόσμος. Δεν υπήρξε ποτέ περικοπή ε, των κονδυλίων για το Εράσμους το αντίθετο μάλιστα. Εμείς ζητούσαμε νέα αύξηση η οποία δεν ε, πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Και ως Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να το λέμε για εκείνους που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, δεν το έχουν ε, ακούσει. Ήταν μια ψευδής είδηση που κυκλοφόρησε. Ναι, ναι, όχι, το συμμερίζομαι. Είπα, Σαμπίν, εξήγησα ότι σε σχέση με την αύξηση που είχε προαναγγελθεί από την Κομισιόν και από τον Άβρατσιτς εδώ για 200 εκατομμύρια γνωρίζαμε ότι τελικά θα γινόταν 100 και μετά τελικά ήταν μόνο 50. Βέβαια όλα αυτά είναι φήμες, δεν είναι επίσημα. Ε, φαίνεται όμως πως η τελευταία είδηση είναι σχετικά βάσιμη. Ε, περνάμε τώρα στο θέμα για το οποίο γίνεται η σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Θέλουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έχουμε ορίσει αυτήν, τη, μάλλον συγκαλέσαμε αυτή τη συνεδρίαση ad hoc για να συζητήσουμε τις τροπολογίες για τη σημαντική αναθεώρηση ε, της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε εισηγήτρια την κυρία Κάμερβέρτε. 950 τροπολογίες υποβλήθηκαν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Ε, μετά από αυτή την ε, σύσκεψη θα πρέπει να ανταλλάξουν απόψεις, αφού μάλλον θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, θα πρέπει να δουν τη δυνατότητα εξέβρεση συμφωνιών ή συμβιβαστικών για ορισμένες από αυτές τις τροπολογίες. Βλέπουμε πως ορισμένες έχουν <clears throat> παρόμοιο χαρακτήρα, άλλες όχι θα είναι μεγάλο έργο, θα πρέπει να το κάνουν ε, οι συγγητρές με τους σκιώδεις. Σίγουρα λοιπόν θα γίνει προσπάθεια από όλους για να καταφέρουμε να διοργανώσουμε διάφορες επαφές με τους εισηγητές, τους σκιώδες για να φτάσουμε στις συμβαστικές. Η πρώτη εξ αυτών των συναντήσεων έχει διοργανωθεί για τις 29 Νοεμβρίου την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι επιτροπές που έχουν ε, αναλάβει την εκπόνηση γνωμοδότηση. εργάζονται από αυτόν. Η ΙΜΚΟ θα δώσει στις 5, η Γιούρη και η ΕΝΒΙ στις 12 Ιανουαρίου, η ΛΥΜΠΕ στις 30 Ιανουαρίου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε τις νομοδοτήσεις και τις ΛΥΜΠΕ που είναι η τελευταία, ώστε μετά να Περάσουμε στην τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτισμού υπό το φως και αυτών των γνωμοδοτήσεων. Αποφασίσαμε λοιπόν η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 28 ε, Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Πολιτισμού. Εύχομαι και είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε στενά σε πνεύμα Αγαστή συνεργασίας. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές απόψεις, το γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά εύχομαι ότι θα να καταφέρουμε από πλευρά των εισηγητών και των σκιωδών να ε, γίνουν όλες οι προσπάθειες για να ε, μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις διάφορες ε, προτάσεις και να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα. Θα θέλαμε να επιτευχθεί συμφωνία υπό την Μαλτέζικη Προεδρία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτή ήταν ο σκοπό των εισηγητριών και 23 Μαΐου να εγκριθεί η γενική προσέγγιση. Θέλω να συγχαρώ τις εισηγήτρες ήδη γιατί ήταν πάρα πολύ δεσμευτική η εργασία αυτή. Αφιερώθηκαν μέρες και ίσως και νύχτες για να μπορέσουμε να δούμε την προκαταρτική εξέταση, την επαλήθευση της νομικής ε, ορολογίας κτλ. κτλ. Δεν ήταν καθόλου απλό, ωστόσο πιστεύω πως θα καταφέρουμε να φτάσουμε τις προθεσμίες και να επιτύχουμε το στόχο μας. Γι' αυτό θα δώσω αμέσω το λόγο τώρα στις δύο εισηγήτρες και μετά στους ε, σκιώδες. Και μετά λοιπόν στους υπόλοιπους. Πρώτα λοιπόν η κυρία Φερχάιεν και μετά η Πέτρα, όχι πρώτα η Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε συμφωνήσει να αρχίσω εγώ και στη συνέχεια η Σαμπίνε να συμπληρώσει. Ε, το είπατε κι εσείς είναι πάρα πολλές οι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Τέτοιου τόμους συνήθω τους ξέρουμε μόνο σε επιτροπέ τύπου ΛΥΜΠΕ και ΙΜΚΟ και όχι απαραίτητο από την Επιτροπή Πολιτισμού. Αλλά αυτό δείχνει ότι η νομοθεσία αυτή και η έκθεση αυτή συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. 950 τροπολογίες συν τις δικές μας που είχαμε υποβάλει εμείς οι συγγήτρες, σύνολο πάνω από 100.000 253 τροπολογίες 253 μόνο για τις αιτιολογικές σκέψεις ε, κατατέθηκαν. Και θέλω να πω εδώ το εξής. Οποιοςδήποτε ε, έχει ε, ζήσει τριμερή διάλογο για ένα νομοθετικό κείμενο θα διαπιστώσει ότι οι αιτιολογικές σκέψεις μετά όλες τις διαπραγματεύσεις συνοψίζονται σε τεχνικές συνεδριάσεις και για μας μας έχει πει η Γραμματεία πολλές φορές ότι υπάρχουν τέτοιου είδους τεχνικές ε, συναντήσεις και παρακαλώ όλους εκείνους που μπήκαν σε αυτόν τον κόπο τον τεράστιο να κάνουν τροπολογίες για τις αιτιολογικές ε, σκέψεις να μην πικραθούν και να μην λυπηθούν εάν δεν βρουν ε, και την κάθε υπό παράγραφο δική τους ας πούμε στο τελικό κείμενο. Προσπαθούμε εκ των προτέρων τις τροπολογίες αυτές να τις εντάξουμε και να τις συνενώσουμε σε λογικούς συμβιβασμούς, ιδιαίτερα για τον εξή και μόνο λόγο, για να έχουμε ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου και στις τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις, για να μην χάσουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, να μην δυσκολέψουμε τη ζωή μας την ίδια, ε, για να μην επιβαρύνουμε πάρα πολύ το κείμενο. Επί της ουσίας θέλω να μπω σε μερικά σημεία. Αρχίζω από τον ορισμό. Τι είστε οπτικοακουστική υπηρεσία στο media. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που προτιμούν την παλιά οδηγία και τον παλιό ορισμό. Αλλά θα ήθελα να πω εγώ εδώ ότι έχει μεταξελιχθεί και λόγω της τεχνολογίας και λόγω της νομολογίας ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είμαστε υποχρεωμένοι και ως νομοθέτες και ως κοινοβούλιο να τα σεβόμαστε αυτά. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχει αλλάξει και ο ορισμός. Υπάρχουν και άλλες επιθυμίες να διευρυνθεί ο ορισμός και να μπει στο... Και, να μπουν και άλλα στο πεδίο εφαρμογής. Ας πούμε, κάποια αλγόριθμοι συντακτικού χαρακτήρα, εκδοτικού χαρακτήρα ή κάποια στοιχεία που είναι σε μια σελίδα του Facebook να εντάσσονται στην οδηγία αυτή. Οι επιθυμίες αυτές μπορεί να είναι κατανοητές, δεν αντιλέγω, αλλά τελικά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα βάλουμε στο πεδίο εφαρμογής και πώς θα ε, ξεχυλώσουμε τρόπο την τον ε, ορισμό. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτή η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών οπτικοκουστικών μέσων και δεν είναι πράγμα το ιδανικό μέσον για να λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Και προσοχή μην την παραφορτώσουμε γιατί θα ε, είναι φρούδες ελπίδες και θα απογοητευτεί ο κόσμος. Και τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν. Και επίση η οδηγία να κρατήσει και μερικά χρόνια, όχι να ξανάρθουμε σε δύο-τρία χρόνια για να ε, κάνουμε σκέψεις για την αναθεώρηση της οδηγίας, γιατί θα μας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις και οι περιστάσεις. Πρέπει και κάπου να διατηρούμε μια ισορροπία. Τι μπορεί από τη μια να κάνει και να προσφέρει οδηγία και από την άλλη να προσπαθήσουμε κάπως να την θωρακίσουμε και για το μέλλον για να μπορέσει να έχει μια λογική ισχύ χρονικά εννοώ. Επίση, τι γίνεται με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και πώ σχετίζεται η παρούσα με εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να την αφισβητήσουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ευθύνε εκείνων που ε, λειτουργούν μια πλατφόρμα εμπορική. Και θα πρέπει ενδεχομένω κάποια σημεία να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε ε, να τα ξεκαθαρίσουμε γιατί καταλαβαίνουμε από τις τροπολογίες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι και αγωνίες. Ότι ενδεχομένω η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο να θυγεί ή να δεν ξέρω, ε, υπονομευθεί κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, γίνεται λόγος ε, για ε, περιεχόμενο βίντεο, για πλατφόρμες ε, παραγωγής ε, βίντεο και ποιος ελέγχει το περιεχόμενο αυτό. Και τι γίνεται και πάλι με τους αλγορίθμους αυτές τις πλατφόρμες και στην οργάνωση και την διάδοση περιεχομένου. Και αυτό έχει σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή όχι. Και υπάρχουν και κάποια live stream που παρέχονται με πλατφόρμες βίντεο θα ε, ε, ενταχθούν σε αυτή την έκθεση ή όχι, σε αυτή την οδηγία δηλαδή. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους κοιόδες ηγητές άλλη μια φορά. Έχουμε πολλές τροπολογίες για την άρση των φραγμών και των εμποδίων. Μέχρι την αρχική παράγραφο 7 φτάνει αυτό. Από εκεί ξεκινάει μέχρι τη δική μας πρόταση ε, ή ακόμα και πιο ευρείες προτάσεις. θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. χωρίς να επιβαρύνονται πάρα πολύ οι πάροχοι του περιεχομένου, αλλά να ανταποκρίνονται στις ε, ε, υποχρεώσεις τους. Υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε με συμβιβασμούς. Και ε, μια άλλη συζήτηση που γίνεται είναι τι γίνεται με τα τυχερά παίγνια. Ε, μπαίνουν ε, στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, δηλαδή ο ηλεκτρονικό τζόγο, και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε σε βάθο στη συνάντηση των σχεδόν. Είχαμε προτείνει μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά με όλες αυτές τις τροπολογίες φαίνεται ότι οι συνάδελφοι συμφωνούν με τη γενική δομική διαρθρωμένη αλλαγή. Προστασία ανηλίκων, προστασία παιδιών επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί, ζητούν κάποιοι, ακόμα περισσότερο. Και υπάρχει και μια σειρά τροπολογιών για τη διαφήμιση, το sponsoring και την τοποθέτηση προϊόντων να μην είναι σε παρέθεση αυτά, αλλά να είναι πριν την παρένθεση. Εμείς θέλουμε να ισχύουν ε, οι ίδιες ε, διατάξεις για όλες τις πλατφόρμες και βίντεο και τα λοιπά. Έγινε μια δύσκολη συζήτηση για τις πλατφόρμες ε, video sharing. Ορισμένοι θέλουν να διατηρηθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι και πάρα πολύ ικανοποιητική. Γιατί είναι να μην ενταχθεί αυτό στην νομοθεσία, αλλά να διέπεται από εθελοντικούς ε, κανόνες δεαντολογίας και να μπορέσουν να νομοθετήσουν τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που χρειαστεί και δεν ε, λειτουργήσει καλά η εθελούσια αυτορύθμιση. Να παραμείνει ανοιχτή αυτή. Είπα για την ε, οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου και για τα θέματα της αστικής ευθύνης. Δεν ξέρω, σε καμία αιτιολογική σκέψη χρειαστεί να τονίσουμε ότι το προνόμιο για την ευθύνη στην οδηγία αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και με καμία μορφή να το περιορίσουμε. υπάρχουν νομικές διαφορές στην αυτόματη επιλογή περιεχομένου ή στη συνειδητή, ε, εσκεμμένη κτλ. Είναι νομικά ζητήματα αυτά. Μετά, εδώ που δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα είναι ε, η διαφήμιση. Ε, για τη γραμμική, επιγραμμική τηλεόραση υπάρχουν γενικές τροπολογίες για η διαφήμιση, 12 λεπτά την ώρα προτείνουν οι περισσότεροι. Σκεφτείτε παρακαλώ και πάλι ότι εμείς ως Κοινοβούλιο τρεις φορές ήδη έχουμε ασχοληθεί. Τελευταία φορά φέτος το Γενάρη το Φλεβάρι, τότε που είχαμε μια μεγάλη έκθεση για την ψηφιακή εσωτερική αγορά, που ορίσαμε και αυτό το θέμα. Τρεις φορές λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία ότι θέλουμε ελαστικοποίηση ε, των προδιαγραφών για την ποσότητα των διαφημίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό που δεν ήταν μόνο του Κοινοβουλίου, ήταν και των κρατών μελών. Και δεν έχω βεβαιωθεί ότι βοηθάει αυτό ε, για την αξιοπιστία μας. Όταν λέμε ελαστικοποίηση και μετά όταν ερχόμαστε στα συγκεκριμένα λέμε καλά, ε, δεν το εννοούσαμε έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι αρνητικό να ε, υποχωρήσουμε εδώ. Αλλά έχουν γίνει πολλές τροπολογίες για τη διαφήμιση και έχω την αίσθηση ότι είναι καλό να έχουμε δύο ε, διακοπές για τηλεοπτικά ε, σποτ, διαφημιστικά. Κάπου στο τέλος πιστεύω να τα βρούμε. θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για θέματα διαφήμισης, για προϊόντα και τρόφιμα κυρίως που περιέχουν ζάχαρη και λιπαρά. Θα δούμε τι θα μας προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και προστασία του Καταναλωτού και πώς θα το κάνουμε, ε, πώς θα τα συγκεράσουμε αυτά με εμφιστάμενες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Τα ίδια ισχύουν. Α, Κάτι άλλο σημαντικό που ξέχασα. Για τα ευρωπαϊκά έργα. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα αυτό. Από το μηδέν ποσόστοση προτείνουν κάποιοι μέχρι 50% για ευρωπαϊκά έργα, ευρωπαϊκές παραγωγές. Ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ορίζουν για πλατφόρμες βίντεο πόσο θα διαρκούν μέχρι. Αν θα προτιμώνται ή όχι οι ευρωπαϊκές παραγωγές, αυτό χωράει συζήτηση, ε, αλλά θα βρούμε κάποιο συμβασμό. Δηλαδή από το 0 μέχρι τα μισά έργα να είναι ευρωπαϊκά ε, υπάρχει και μεγάλο περιθώριο συμβιβασμού. Για την ακαιρεότητα του σήματος νομίζουμε ότι οι δικές μας προτάσεις είναι οι καλύτερες και αξίζει να υποστηριχθούν. Θα σταματήσω εδώ. Έχουμε δύο συναντήσεις των σκιωδών προβλέψει. Πρώτη είναι στις 29 του μηνός και η δεύτερη στις 12 Ιανουαρίου, 9 με 11 κάθε φορά. Στην πρώτη συνεδρίαση δεν έχουμε διερμηνία, τουλάχιστον θα φροντίσουμε στη δεύτερη να έχουμε. Γιατί είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα και σύνθετο, ώστε χωρίς διερμηνία να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Αλλά με αυτές τις δύο συνεδριάσεις νομίζω σχεδόν δεν θα τελειώσουμε, δεν μας φτάνει. Γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η οποία θα αποφασίσει μόλις στις 30 Ιανουαρίου. Και όλα τα επίμαχα θέματα και τα θέματα της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών θα τα βρούμε μπροστά μας. Μπορεί να είδατε ότι και στις δικές μας τροπολογίες Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές και κάποιες βελτιώσεις. Και στην ε, ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος και μας. Θέλουμε να είναι και θέλουμε και να ορίζεται αυτό στην νομοθεσία. Υπάρχουν τροπολογίες που λέγουν καλή ιδέα και συμφωνούμε <laughs> αλλά η ακαιρεότητα και, και η ανεξαρτησία είναι κάτι που θα πρέπει να το ξέρουν και οι κυβερνήσεις και να το σέβονται. Αυτά και σταματώ εδώ προς το παρόν. Πέτρα, ευχαριστώ. Μια μεγάλη επισκόπηση μας έκανες. Για κάποια σημεία έχουμε αποκλήσεις ενώ για κάποια άλλα υπάρχουν συγκλίνωσες προτάσεις και ελπίζω τέλο πάντων να βρούμε μια ισορροπία μέσω διαλόγου. Η Σαμπίνα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ και την Πέτρα που έδωσε μια ευρύτατη επισκόπηση των τροπολογιών, τουλάχιστον της δικής μας Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Οι άλλες ε, επιτροπές ακόμα το συζητούν. Έχουμε επαφές μαζί τους σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. Γνωρίζω ότι το συζητάνε οι ομάδες και στο στάδιο της ε, εκπόνησης των ε, τροπολογιών. Προσπαθούμε να είμαστε σε στενή συνεργασία από την αρχή με τις γνωμοδοτούσες επιτροπές ε, για να τα βρούμε. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες είπαμε και μάλιστα πάρα πολύ διαφορετικές θέσεις και απόψεις για τα επιμέρους θέματα. Τα είπε η Πέτρα Δηλαδή, μερικές είναι η μέρα με τη νύχτα. Για την ελαστικοποίηση ή για την ε, αυστηροποίηση ε, της οδηγίας για τις ε, διαφημίσεις. Υπάρχουν προτάσεις που απέχουν πάρα πολύ. Άλλοι ζητούν την πλήρη αυστηροποίηση και άλλοι την πλήρη απελευθέρωση. Πρέπει να βρούμε μία λύση έτσι ώστε όλοι οι ε, ενεχόμενοι να έχουν ε, δίκαιους και ίσους ε, κανόνες παιχνιδιού στο μέλλον. Γιατί συγκλίνουν τώρα τα μίντια, δεν έχουμε τη διάκριση του παρελθόντος που ξέραμε ποιο μέσο είναι ποιο. Τώρα όλα είναι ένα περίπου και στο μέλλον θα έχουν περισσότερη συνένωση. Και θα πρέπει να προστατεύουμε και τους ε, ε, ανήλικους και τα παιδιά. Πρέπει να γίνει λοιπόν μεγάλη συζήτηση για τις πλατφόρμες video sharing. Και πρέπει να δούμε ποια ε, θέματα τα ρυθμίζει η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει αστική ευθύνη ο πάροχος. Και με την οδηγία αυτή για τα οπτικοακουστικά δεν μπορούμε να καταργήσουμε την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, άρα πρέπει να βρούμε λογικές λύσεις για καλύτερη προστασία πάντα και των παιδιών και των ανηλίκων, αλλά γενικότερα και των καταναλωτών. Χωρίς να υπονομεύεται η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάντως ε, σίγουρα θα καταλήξουμε σε λογικό συμβιβασμό. Για το θέμα έργα, πρέπει να σας πω ότι δεν θέλαμε εμείς να την αποδυναμώσουμε, αλλά να τη βοηθήσουμε. Δηλαδή, να μην έχουμε μια υπερρυθμιστική αρχή στην Ευρώπη, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω είχε τέτοια πρόθεση να έχουμε έναν υπερφορέα δηλαδή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με βάση το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ και των συμβάσεων και των συνθήκων που έχουμε έχει αυξημένη ευθύνη και ε, πρέπει να ρυθμίζεται αυτό και με την σύγκληση και με τις διασυνοριακές προσφορές και παροχές περιεχομένου που αυξάνονται ε, πρέπει να υπάρξει σχετική ρύθμιση για την έργα και μπαίνει και ένα ε, ζήτημα όχι μόνο πολιτικό αλλά και τεχνικό. Και θα πρέπει να ακούμε και τους εκπροσώπους των κρατών μελών και τους πολιτικούς αλλά και τους ειδικού, τεχνικούς εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με θέματα εφαρμογής και ελέγχου. Και αυτός ο Ευρωπαίος ε, συντονιστής το γκρουπ αυτό των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών έχει συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει και θα δούμε τι χρειάζεται να αλλάξει και τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεσή μας. Για την ανεξάρτητη ε, ρυθμιστική αρχή τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια Όλοι στο Κοινοβούλιο θελήσαμε στα κράτη-μέλη η εποπτεία των μίντια να είναι τελείως ανεξάρτητη. Οι δομές, το πώς θα το κάνει η κάθε κυβέρνηση ε, ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή, ε, όχι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης και κάποια θέματα που λειτουργούν σωστά δεν θα πρέπει να καταστραφούν τελείως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει λειτουργική ανεξαρτησία του ρυθμιστεί ας πούμε, του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ε, από το κράτος. Από την κυβέρνηση θα πρέπει να είναι διακριτός ο ρόλος και ε, επίσημα. Και τέλος θα βρούμε κάποια λύση. Σε ένα άλλο θέμα που ε, αναφέρουν και οι τροπολογίες είναι πώς απολύονται ή πώς πάβονται τα μέλη ενός Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει με διαφάνεια ε, Και γιατί καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πράγματα μονοπλευρά, μονομερή, που δεν συνάδουν με την εργατική νομοθεσία και ε, ε, αφήνουν περιθώριο για αυθαιρεσίες. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο πάυσης ή απόλυσης. Υπάρχουν και κάποιες θητείες που λήγουν, κάποιες συμβόλαια που λήγουν και μετά υπάρχει ο κίνδυνος να βάζει εκλεκτούς της κάθε κυβέρνηση. Αυτό παύση η βάση των θεμάτων, πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Επίσης η πρόθεση των ευρωπαϊκών παραγωγών, των ευρωπαϊκών έργων και πάλι ορισμένοι δεν θέλουν καθόλου, άλλοι θέλουν τα μισά να είναι ευρωπαϊκά. Εμείς στο κάτω-κάτω είμαστε Επιτροπή Πολιτισμού και μας πέφτει λόγος και είναι και ευθύνη μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προάγει ε, την ποικιλομορφία και την πολιτισμική και τη μηντιακή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση και με χαρά περιμένω τη συζητήση με τους κοιόδες συγητές. Αλλά είδαμε από τις τροπολογίες ότι και στο εσωτερικό κόμμα των πολιτικών ομάδων υπάρχει ε, μεγάλη ανάγκη συζήτησης. Υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες και διχογνωμίες στο εσωτερικό της ίδιας πολιτικής ομάδας. Το βλέπουμε από τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πράγματι. Σωστό αυτό. Να πούμε ότι χρειάζεται βάθυνση. Αλλά υπάρχει βούληση και είμαι σίγουρη ότι θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα δώσω το λόγο σε αυτούς που το ζήτησαν Λιουερ, Τόμ και Τρούπερ μετά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι. Γραμματικά και επίσης. Αντρέ Παρκαλό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλησπέρα. Συγγνώμη που έλαβα το λόγο αλλά πρέπει να φύγω και θα ακούσω όλους τους συναδέλφους. Πάντως, οι συνεργάτες μου θα σημειώσουν αυτά που θα πούν οι συνάδελφοι. Θα περιοριστώ λοιπόν σε δύο κυρία ζητήματα από το σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες που λάβαμε. Δηλαδή, εκτός από τις ποσοστώσεις και δασμούς, όπου έχω ξεκάθαρες αντιρρήσεις, επειδή έχουμε ευρύτερα ζητήματα που δεν έχω χρόνο τόσο πάντων να αναφέρω στα πλαίσια πάντως της τέχνης του εφικτού. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις πλατφόρμες για το video sharing και την επιλογή της εισηγήτριας να περιλάβει αυτές νέες σχετικά επι, επι, υπηρεσίες μάλλον στο πεδίο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή επιθυμητό. Πάντω κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν ήδη για τη δυνατότητα ευελιξία οπότε προσβλέπω σε περαιτέρω διερεύνηση. Η ECR συμφωνεί με τους στόχους της Επιτροπής για την ενίσχυση των στόχων που αφορούν ιδιαίτερα τους ανηλίκους. Γι' αυτό ακριβώς συμφωνούμε με αυτά που θέλει η Επιτροπή για την διεύρυνση δηλαδή του πεδίου σε σχέση με πλατφόρμες video sharing σύμφωνα με τις τροπολογίες μας. Πρέπει επίσης να υπάρχει και μια προσέγγιση συντεριθμιστική ώστε να αποφύγουμε υπερβολικές απαιτήσει εθνικές για τη βιομηχανία προστατεύοντας ταυτόχρονα βέβαια και τους ανήλικους online. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας κίνδυνος στις προτάσεις. Δηλαδή οι προτάσεις φαίνεται να υπολείπονται εδώ. Δηλαδή, καταρχάς, διευρύνουν τους κανονισμούς όσον αφορά τι εμπορικές επικοινωνίες στα VSPs. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εδώ έχουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένη ευθύνη όσον αφορά τη διαφήμιση. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που το καταδεικνύουν αυτό. Επίσης έχουμε και μία πρώτερη γνώση του περιεχομένου το οποίο δεν ισχύει πάντοτε στην πράξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχουμε τοποθέτηση προϊόντων. Αυτές λοιπόν οι διαφορές θα πρέπει να προσδιοριστούν σε οποιαδήποτε πρόταση πριν η ECR λάβει υπόψη τη οποιασδήποτε επέκταση του διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή για τα VCR ε, και σε, και σε σχέση με τον κανονισμό για τις υπηρεσίε τη υπηρεσία Να πω επίσης ότι για τους VSPs πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα προελέχου του περιεχομένου και ο έλεγχος, ο συγκεκριμένος έλεγχος του περιεχομένου δεν θέλουμε να οδηγήσει σε μορφές λογοκρισίας. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχει μια κατάσταση όπου οι πολίτες σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης δεν θα μπορούν να ανεβάζουν τα βίντεο τους στο ίντερνετ αφού έχουν ελεγχθεί, τέλο πάντων από κάποιον στο περιεχόμενο. Μετά, οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν και με τις ε, αρμοδιότητες της, της οδηγίας για το εμπόριο που αφορούν την ανάπτυξη ολόκληρης της πλατφόρμας της εμπορικής online της βιομηχανίας αυτής. Θέλουμε λοιπόν να διατηρηθούν παραπομπές στην οδηγία στα 14 και 15 όπως κάνει η συγγήτρια και αυτό είναι νομίζω χρήσιμο όσον αφορά την προστασία. Όμως η προστασία αυτή δεν φτάνει όταν μιλάμε για την ευθύνη των VSPs κάτι το οποίο νομίζω θα οδηγήσει στην κατάρρευση της οδηγίας. Δηλαδή όταν ζητάμε από τους VSPs να προελέξουν το περιεχόμενο τότε τι γίνεται, ποιο είναι το επόμενο βήμα, πώς εφαρμόζονται όλα αυτά πούμε, στα πνευματικά δικαιώματα στην τρομοκρατία α πούμε. Τέλος, αυτή η προαπέτηση για τους VSPs δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά, δηλαδή περιεχόμενο το οποίο φορτώνεται αναδευτερόρθω σε μεγάλους όγκους. Ε, πώς μπορούν να το καλύψουν όλο οι VSPs και με τι επιπτώσεις και πώς αυτό θα έχει επιπτώσει σε μικρές βυσπίσεις ή σε startups. Γι' αυτό ακριβώς έλεγα ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές χάρη αλλαγών, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Όταν κάνουμε αλλαγές, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν τεκμήρια για αυτές τις αλλαγές και θα πρέπει να παρέχουν σαφήνεια νομική, γιατί οι αλλαγές αυτές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε παράπλευρες ε, απώλειες. Να το έχουν αυτό λοιπόν υπόψη τους ε, οι συνάδελφοι όταν θα έχουμε τις επόμενες συνεδρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η συνάδελφο, ο, ο λόγος συνάδελφο Τόμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι μόλις έρχομαι από μια συνεδρίαση όπου η φιλελεύθερη ομάδα ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και προβληματίζεται. υπάρχει πολλοί κόσμος που αναρωτιέται ποια θα είναι η θέση μας και πώς θα αποκρισταλωθεί αυτή. Ε, χτες το βράδυ κοιμήθηκα μόνο τρεις ώρες γιατί έπρεπε να ξυπνήσω νυχτιάτικα να τρέχω στο αεροδρόμιο. Και ξέρετε ότι και αυτές τις τρεις ώρες που κοιμήθηκα Έβλεπα στον ύπνο μου τις συζυγήτριες και την οδηγία. Λοιπόν, για να μην συνεχίσετε και με βλέπετε και εσείς και έχετε εφιάλτες, ε, θα τα πω ε, στα αγγλικά, γιατί όταν μιλάω στον έχω την αίσθηση ότι δεν με καταλαβαίνετε όλοι. Για να μην σας χαλάσω και τον ύπνο. Θα μιλήσω ευρωγλώσσα τώρα, θα με καταλάβετε ελπίζω. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει κάποια καλά πράγματα όπως οι απαιτήσει για την υποθέτηση των προϊόντων, η προστασία των ανηλίκων, ιδιαίτερα στο video on demand και η υποχρέωση των χωρών μελών να καθορίσουν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιες διατάξεις κατά την άποψή μας πρέπει να αφαιρεθούν. Μία από αυτές αφορά τις ποσοστώσεις. έχουμε ένα ποσοστό από 1 μέχρι 50. Έχουμε αυτές τις υπηρεσίε on demand. Οι συνεισηγήτριες Πέρα να βγάλω τα ακουστικά μου γιατί ακούω τη μετάφραση λέει η ομιλήτρια. Λένε 30 του. Αυξάνουν. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε του πολίτε να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι υπηρεσίε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ποσοστώσεις βοηθάνε σε αυτό. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να συμπληρώσουμε το με εθνικά έργα. Για να δω, εδώ, αναρτημίσω και τον ήχο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμπληρώσουμε το κατάλογο με εθνικά έργα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εδώ μπορούμε να προωθήσουμε ευρωπαϊκά έργα άλλων χωρών δηλαδή. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό στα πλαίσια των υπηρεσιών on demand που βεβαίως ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αγοράς φτηνών ευρωπαϊκών προϊόντων για να συμπληρωθούν κατάλογοι. Θα πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά έργα, οι ευρωπαϊκέ δημιουργίε να φαίνονται κάπω έτσι μεγαλύτερε και αυτό μπορεί να γίνει φαντάζομαι με τεχνητό τρόπο. Πάντω ο στόχο τη πρόθεση των ευρωπαϊκών έργων δεν νομίζω να επιτευχθεί και θα υποφέρουν οι κατανότε από αυτό. Μετά εδασμοί. Η θέσπιση οικονομική συμβολής νομίζω προκαλεί ανησυχίε. Η Κομισιόν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα αυτή των χωρών μελών να ζητήσουν τα on demand για να συμβάλλει και προ τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων. Υπάρχει όμως μια δικαιοδοσία εδώ. Τι γίνεται και ποιε αρμοδιότητε έχουμε. Γιατί εδώ θα έχουμε μια ανεπιθύμητη κατάσταση όπου αυτοί που παρέχουν αυτέ τι υπηρεσίε on demand σε όλε τι 28 χώρε μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν σε 28 διαφορετικά εθνικά ταμεία για τι πλατφόρμε. Οι πλατφόρμες να είναι υπεύθυνε για κάθε βίντεο το οποίο ανεβαίνει σε αυτέ τι πλατφόρμε. Δεν ξέρω, εδώ χρειάζεται πλήρη εποπτεία Απόλυτο monitoring δηλαδή, λέω μιλήτρια. Τώρα για το βλαβερό περιεχόμενο, επιλαβές. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο βέβαια αυτό το περιεχόμενο είναι βλαβερό ή όχι. Πλαίσιο, νομικό. Τι γίνεται με αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ της μέγιστης ε, εναρμόνισης για τους ε, κανόνες που αφορούν το περιεχόμενο. Συνεπώς, Θέλουμε να υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία για το έργα. Δεν θέλουμε ο ρόλος του να είναι χαμηλότερος, λιγότερος. Θέλουμε να αναγίνεται αναφορά στην οδηγία, όμως θα θέλαμε να μην σημειωθούν εδώ καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε ανοιχτοί σχετικά με το πόσο λεπτομερής πρέπει να είναι παράγραφη για αυτό το θέμα. Οπότε θα θέλαμε να περιμέναμε και την νομοδότηση ΣΥΝΚΟ. Αυτά περίπου είχα να πω εγώ. Νο... Νομίζω είχαμε γύρω στις 100 και βάλε τροπολογίες για αυτά τα θέματα. Θα μπορώ να σας απαριθμίσω αν σας αρέσει, αλλά όχι δεν θα το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, που δεν το κάνατε λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ γιατί θα ανησυχούσαμε. Τώρα θα δώσω το λόγο λέει η Πρόεδρος στην συνάδελφο Τρούπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις εισηγήτριές μας για την παρουσίαση αυτή και τους υπολείπους ε, που μίλησαν από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Να αρχίσω με την πρόταση για τη δομή της οδηγίας και της τροπολογίας ε, να μπουν τόσα πολλά ε, εκτός παρενθέσεως. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τους λόγους της να επιλέξει αυτή την προσέγγιση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος εξάντε ε, και για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα πρέπει να φυγεί η αντίστοιχη οδηγία. Διότι αυτό πρόκειται ε, εδώ για ένα παθητικό ρόλο διαβιβαστεί απλώς του περιεχομένου της πλατφόρμας και δεν ξέρουν οι ψηφιακοί ε, χρήστες και πάροχοι ε, ποιο είναι το περιεχόμενο. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που οι πλατφόρμες δεν έχουν μόνο παθητικό ρόλο αλλά και ενεργητικό και εμπορικό. Βγάζουν καταλόγους, πουλάνε ε, το περιεχόμενο το οργανώνουν και το παρέχουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι παθητικός ο ρόλος τους μόνο, έχει γίνει ενεργητικός και πρωταγωνιστικός. Παρ' όλα αυτά λέμε να μην αλλάξουμε τη βάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά αυτό που θέλουμε είναι διευκρίνηση για το παθητικό και το ενεργητικό, τι εννοούμε κάθε φορά. Χρειάζεται σαφής ορισμός για αυτό το σκοπό. Επανέρχομαι τώρα στη δομή της οδηγίας, γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ όσων γνωρίζω εγώ και καταλαβαίνω, υπάρχουν περιεχόμενα σε πλατφόρμες που είναι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και χρειάζονται πιο ισχυρή ρύθμιση από ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αλλά υπάρχει και περιεχόμενο το οποίο ε, έχουν ε, παραγάγει οι ίδιοι χρήστε, ε, user user-generated ε, content λέγεται αυτό, το οποίο δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα και μπορεί να κυκλοφορεί από χρήστη σε χρήστη. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος ε, της ομάδας των ρυθμιστικών αρχών, έργα. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και εδώ και πάλι αυτά τα βασικά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σωστά. Ότι ναι, θέλουμε, χρειαζόμαστε τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο και στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουν πιο ενισχυμένη συνεργασία σε καμία περίπτωση να μην συμμετέχουν στην νομοθεσία, απλώς να εποπτεύουν, να παρακολουθούν την εφαρμογή της οδηγίας στη μεταφορά με καλή ανταλλαγή μεταξύ τους και οι κοινέ αξίες και αρχές και τα πρότυπα που συμφωνήσαμε να βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί ξέρουμε όπου ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες ε, με αρνητικές εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Δεν θέλει καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τραβήξει στο μέρος τις περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά να υπάρχει δίκαιη ρύθμιση του μηδιακού τοπίου. φαίνεται ένα συμβιβασμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει προθυμία να βρεθεί μια διατύπωση που να λέει ότι είναι ανεξάρτητες οι ρυθμιστικές αρχές από την κυβέρνηση και κρατικές δομές. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έρχομαι τώρα εκεί που χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις. Λοιπόν, κάτι που θεωρώ σωστό καταρχήν. Οι πλατφόρμες video sharing να είναι περισσότερο στο πεδίο της ευθύνη ιδιαίτερα για την παροχή ποιοτική διαφήμισης. Ήταν και δική μου πρόταση αυτή. Αλλά δεν συμφωνώ με την ποσοτική ρύθμιση για την επιγραμμική τηλεόραση. Ε, να απελευθερωθεί δηλαδή η παροχή των διαφημίσεων. Αν κοιτάξω το τηλεοπτικό τοπίο και αυτό που θέλουν πολλοί καταναλωτές είναι να μην διονγκωθεί υπερβολικά ο χρόνος που αφιερώνεται στη διαφήμιση. Να παραμείνουμε στο 20% την ώρα. Το εν πέμπτο, δηλαδή 12 λεπτά. Διαφωνώ με τους φιλελευθέρους για τα ευρωπαϊκά έργα, για την πολιτιστική ποικιλομορφία, τις ευρωπαϊκές παραγωγές και δημιουργίες. Εγώ θέλω να έχουμε κάποια ποσόστοση για ευρωπαϊκά έργα και με το επιχείρημα της αγοράς που λέει υπάρχουν πλατφόρμες για video on demand. Μα πρέπει να το κάνουν γιατί ο κόσμος το θέλει. Όταν θέλεις να έχεις ένα ελκυστικό πακέτο στην προσφορά σου πρέπει να έχει και ευρωπαϊκό περιεχόμενο και νομίζω το κάνουν ήδη. Ε, Τη τάξη του 20, 25 και 27% είναι η προσφορά των ευρωπαϊκών δημιουργιών και παραγωγών. Βεβαίω και να γίνεται, γιατί εμεί θέλουμε να το έχουμε αυτό σε Επιτροπή Πολιτισμού και να είναι και πιο ορατή και πιο προβεβλημένη η ευρωπαϊκή παραγωγή. Άρα κάντε το 30%. Ακούστηκε και μια άλλη ιδέα για τους συναδέλφους για τα social media, να μπουν και αυτά στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα θέματα αυτά τα ενεργητικά και παθητικά. Τι ρόλο έχει ο πάροχος. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα τυχερά παιχνίδια εδώ. Προστασία των ελίκων προφανώς και σωστό, αλλά θέλω να το ρυθμίσουμε και με τρόπο πολύ σαφή, πιο σαφή από ό,τι προτείνεται εδώ. Για το sponsoring και για την τοποθέτηση προϊόντος και δεν θέλω σε καμία περίπτωση σε παιδικές εκπομπές να έχουμε διαφημίσεις και ότι θέλω να αποδυναμωθεί αυτό το όριο που έχουμε τώρα ότι η διακοπή για διαφήμιση θα γίνεται κάθε μισή ώρα, όχι πιο νωρίς. Η ακαιρεότητα του σήματο βεβαίω να παραμείνει και να διαφυλαχθεί και θέλω τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, έχουν κανόνες και επίσης το θέμα της πρόσβασης ε, για τους αναπήρους να μην είναι στη Γενική Οδηγία και την πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. Το ζητούν και οργανώσεις τους τον ΑΜΕΑ να ενταχθεί στην παρούσα οδηγία. Και σε ό,τι αφορά τη συν ε, νομοθεσία, ρύθμιση, όταν δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες να ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν και σε νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή να υπάρχει μια πολιτική παρουσία καθοδήγηση της πολιτείας και να μην είναι απολύτως εθελοντικό το σύστημα, δεντολογία δηλαδή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει πάντα να είναι χωριστή διαφήμιση από το περιεχόμενο του ουσιαστικό και όταν πρόκειται για τοποθέτηση προϊόντος να το λέει και να μην είναι γκρίζα διαφήμιση ή υποβολημία. Αυτά, κάποια άλλα θέματα εχνηλασιμότητας, ανιχνευσιμότητας. Σταματώ αυτή τη στιγμή εδώ, σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, ο συνάδελφος Βέντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τις συναδέλφους που εκπώνησαν αυτό το σχέδιο έκθεσης για την πολύ σκληρή τους δουλειά. Ε, και οι συμβιβαστικές ε, θα απαιτήσουν πολύ δουλειά. Λοιπόν, το άρθρο 35 δεν είναι πολύ σαφές. Είναι αυτό που κάνει λόγο για τους ε, διορισμούς στα αριθμιστικά όργανα. Η Κομισιόν κάνει λόγο για ε, προστασία από αυθαίρετες ε, παρεμβάσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Το να αφαιρεθούν οι παράγραφοι αυτοί από το άρθρο 35 μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση στο επίπεδο των κρατών μελών όσον αφορά τις ε, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά τη χώρα μου. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικά. Δεύτερο θέμα γίνεται αναφορά στην διαφημίμηση και στις ώρες. Το να αλλάξουν τα όρια τα καθημερινά μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική εμπορευματοποίηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων και υπερβολική παρουσία διαφημίσεων σε συγκεκριμένα ωράρια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της αξίας του χρόνου διαφήμισης και την μείωση της αξίας του εισμεμονωμένης διαφήμισης. Οι θεατές μπορεί να πάψουν να παρακολουθούν τα παραδοσιακά μέσα λόγω αυτής τις υπερβολικής διαφήμισης. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια λύση που θα προστατεύσει τους καταναλωτές και κυρίως τους ανήλικους θεατές. Επίσης, οι τηλεοράσεις χρειάζονται βέβαια τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Ε, γι' αυτό θα πρότεινα το 20% στη διάρκεια της ημέρας, αλλά χωρίς να περβαίνουν τα 15 λεπτά την ώρα. Ευχαριστώ. Για την ώρα αυτά. Ο κύριος Γραμματικάκης. Ήξερα, κύριε Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το θέμα, αλλά όταν δει κανένας αυτόν τον όγκο των τεσσάρων εδώ βιβλίων, ολόκληρα βιβλία έχουν γίνει τροπολογίες, πρώτα πρέπει να θαυμάσει και να ευχαριστήσει τις συναδέλφους Πέτρα και Σαμπίνα, εγώ θα μπορούσα να το κάνω όλο αυτό, και δεύτερο να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό. Νομίζω είναι η εποχή αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσες πολλές επιτροπές ανακατεύονται. Νομίζω ότι το θέμα θίγει την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα περιοριστώ πολύ γρήγορα σε τρεις ε, βασικές παρατηρήσεις γιατί η Πέτρα έκανε μια γενική εισαγωγή ε, κατανοητή απολύτως και τη συμπλήρωσε η Σαμπίνα. Ε, πρώτα πρώτα για πρώτη φορά εγώ ασχολήθηκα λιγάκι με το θέμα των διαφημίσεων επειδή είμαστε Επιτροπή Πολιτισμού νομίζω ότι τα 12 λεπτά είναι υπέρα αρκετά πρέπει να δώσουμε τον τόνο εμείς αλλά απ' την άλλη είναι σεβαστό το επιχείρημα νομίζω η Πέτρα το τόνισε ότι δεν μπορούμε να ζητάμε αλλαγές και μετά να ξαπανερχόμαστε στα ίδια. Νομίζω εκεί πολύ εύκολα θα βρεθεί μια λύση Είμαι τελείως αντίθετος με το να ανακατευτούν τα τυχερά παιχνίδια με όλα αυτά. Θα κάνω πιο, πιο πολύπλοκη την πραγματικότητα. Και εγώ θα τονίσω τώρα γιατί ασχολήθηκα ειδικά με τις ρυθμιστικές αρχές. Πρώτα-πρώτα γιατί η Ελλάδα έχει πολύ πικρή πείρα από αυτά. Δεν υπήρξαν ποτέ ουσιαστικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς με τις δικές μου τροπολογίες θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι αρχές θα είναι ανεξάρτητες όχι μόνο στα χαρτιά, που σημαίνει κάποιος νομικός διαχωρισμός, αλλά κυρίως στην πράξη. Γι' αυτό το τονίζω, ζητούμε οι διορισμοί να γίνονται των μελών μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, έχει μεγάλη σημασία, να έχουν συγκεκριμένη θητεία που να μην μπορεί να διακόπτεται Όλα αυτά στηρίζονται σε κακές εμπειρίες των τελευταίων δέκα χρόνων όσο παρακολουθώ αυτά τα ραδιοτηλεοπτικά πράγματα στην Ευρώπη. Επίσης η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι λειτουργική και ανεξάρτητα από την αδυναμία ορισμού ενός ή περισσότερων μελών για οποιοδήποτε λόγο. Εγώ ιδιαίτερη σημασία, αν μου επιτρέπετε και τελειώνω, δίνω στην τροπολογία υπαριθμών 997, καταντάμε να μετράμε μέχρι το 1500, δεν ξέρω που θα φτάσουμε, η οποία ζητά διαφάνεια στο θέμα της χορήγησης και ανανέωσης των αδειών. Δεν θέλουμε προφανώς να πούμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια και οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς. Ειδικά για τους ε, δημοκράτες και σοσιαλιστές τέτοια κριτήρια είναι νομίζω απαραίτητα και το μόνο που έχω να ευχηθώ τελειώνοντας είναι τουλάχιστον στη διάρκεια της δικής μου θητείας, δηλαδή δυόμιση τρία χρόνια έχουμε ακόμα, να δούμε μια πραγματικότητα μέσα από αυτό το χάος, να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα. Υπάρχει αρκετή αισιοδοξία, αλλά χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και εγώ έχω την απόφαση να κάνω από μέρους μου το καλύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συγγητές και τον σύντροφο γραμματική Κάκη. Συμφωνούμε με την έκθεση. και με πολλές πτυχές της πρόθεση ευρωπαϊκών έργων, ευελιξία στη διαφήμιση. Παρ' αυτά θεωρούμε ότι κάποιες αξίες απαιτούν αυστηρή προσέγγιση, προστασία δηλαδή των αλληλίκων και απολογία μίσους. Θεωρούμε ότι αυτό το θέμα με τις πλατφόρμες έχει τεράστια σημασία γιατί ποτέ δεν υπήρξαν τόσες πληροφορίες και τόσο υλικό online και καταναλώνεται αυτό το περιεχόμενο με το ίδιο τρόπο online και αυτοί οι καταναλωτές συνήθως είναι ανήλικοι και δεν διακρίνουν από τα, τα παραδοσιακά, από τα online μέσα. Οπότε είναι πιο ευάλωτοι αυτοί οι καταναλωτές αν δεν υπάρχουν, υπάρχουν συστήματα που τους προστατεύουν. Και νομίζω σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε εμεί περισσότερο στην έκθεσή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζηλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω απλά να επανέλθω σε δύο ζητήματα που τίθενται μέσω αυτή τη οδηγία, που είναι στην ουσία τι πρότυπο επιθυμούμε για τα οπτικοακουστικά μέσα και έπειτα σε ποιου θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνε. Ε, θα ήθελα ε, καταρχά να θέσω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, τι περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τι οπτικοακουστικές Υπηρεσίε. Εγώ πιστεύω ότι περιμένουν ε, περιεχόμενο και περιεχόμενο περισσότερο από ό,τι διακοπές διαφημίσει κάθε 20 λεπτά. Βέβαια οι διαφημίσεις ε, φυσικά αν είναι αλήθεια χρηματοδοτούν το περιεχόμενο και γι' αυτό το λόγο και συμμερίζομαι την ιδέα να στηρίξουμε την ευελιξία που δίνεται στη χορηγία αλλά και για την τοποθέτηση προϊόντων αλλά ε, νομίζω όπως και πολλοί εδώ πιστεύω ότι η αρχή της αυστηρής οριοθέτησης για τα ωράρια είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από το αμερικανικό πρότυπο και που αποτελεί ίσως και έναν από τους πρώτους τους πυλώνες του ευρωπαϊκού μοντέλου σε αυτό το τομέα. Επίσης αυτό που αναμένουμε από τις οπτικοακουστικές μας υπηρεσίες είναι νομίζω να προτάξουν το ευρωπαϊκό περιεχόμενο που συχνά είναι ποιοτικό και αποτελεί λόγο περηφάνειας για πολλούς από εμά και νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πυλώνας του μοντέλου του ευρωπαϊκού που προανέφερα και γι' αυτό θα ήθελα η ποσόστοση για ευρωπαϊκά έργα να εφαρμόζεται και στις ε, υπηρεσίες ε, ε, ε, βίντεο αλλά demand, video on demand κατά 40%. Σαφής λοιπόν περιορισμός των διαφημίσεων είναι οι δικές μου απόψεις και δεύτερον η πολιτιστική ποικιλομορφία μέσω αυτού του, της πρότασης. Το άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι σε ποιον θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες τελικά, για ποιους θα ισχύουν. Εγώ στηρίζω αυτά που προτείνουν οι συγγήτρες, ώστε οι κοινοί κανόνες να ισχύουν για το σύνολο των οπτικοκουστικών μέσων, όποια και αν είναι αυτά. Και πέρα από αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα που αφορά τάσεις που διαπιστώσαμε με ευκαιρία τις Αμερικανικές εκλογές και που επέτρεψαν να παρατηρήσουμε το χώρο που κάλυψαν τα κοινωνικά, καλύπτουν τα κοινωνικά δίκτυα. Σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε, βλέπουμε ότι 44% των Αμερικανών χρησιμοποιούν το Facebook ως πρώτο χώρο ενημέρωσης και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρόσφατης προεκλογικής εκστατείας και μάλιστα το Facebook χάρη σε οπτικοκοστικά περιεχόμενο που προβάλλεται από αυτή την πλατφόρμα και έπειτα είδαμε πως το Facebook έχει υπογράψει νομίζω 140 συμβάσεις με διάφορους Εντάξει. Ε, ε, δίκτυα παροχής ε, περιεχομένου ακριβώς με στόχο να τροποποιηθεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο ώστε να ταιριάζει στο facebook. Έχουμε δηλαδή ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιεί οπτικοακουστικό περιεχόμενο και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της οδηγίας αλλά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγώ υπερασπίζω την ιδέα μιας σαφούς ένταξης των κοινωνικών δικτύων στην οδηγία δεδομένης δεδομένου του εύρους του φαινομένου και της χρήσης των καταναλωτών αυτών των δικτύων. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Σοριντρόβα τώρα. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στις εισηγήτριες ε, πρώτα απ' όλα. Με όλες αυτές τις τροπολογίες πάνω από 150, 950 ναι, ε, συγγνώμη, γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε και τις τροπολογίες των διαφόρων επιτροπών. Πολλή δουλειά λοιπόν ε, έχουν και θέλω να υπογραμμίσω ότι πιστεύω πως υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία. Από τη μια έχουμε την προστασία των ανηλίκων, από το βλαβερό περιεχόμενο έχουμε τον ε, ε υποδάβληση μίσους, και έπειτα έχουμε και τις πλατφόρμες ε, βίντεο sharing. Όλοι υπογράμμισαν την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και άνευ αυτής της ε, ε, κάλυψης δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε την προστασία των ανηλίκων. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου με τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε να μπορούμε μάλλον να προχωρήσουμε σε ελέγχου, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και να αποφύγουμε την υποδάβληση ε, του μίσου ή τη βία, και μάλιστα να ελέγξουμε και το περιεχόμενο των ε, πλατφορμών video sharing ή υπηρεσιών ε, κατά παραγγελία. Ε, εάν ε, επίσης στις διαφημίσεις έχουμε 20% ή 30% που προβλέπονται από την Επιτροπή και από τις εισηγήτριες. Αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει ωστόσο σημασία είναι να υπάρχει περιεχόμενο ευρωπαϊκό. Επίση, μιλήσαμε για το θέμα της προσβασιμότητας, ειδικά για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ε, έχουμε ευθύνη όχι μόνο οι, τα κατημέλη και οι πάροχοι των κατορμελών θα πρέπει να έχουμε μία πρόταση ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει στο σεβασμό αυτών των ευθυνών, συντήρηση στην ανταπόκριση σε αυτές τις ευθύνες πρόκειται για λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις τροπολογίες, ούτως ώστε η Κομισιόν να βοηθήσει τα κρατημέλη να ανταποκριθούν σε αυτή του τη ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ ε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριες ε, και για τις εισηγήσεις τους τις απόψινές ε, και για τα θέματα τα οποία μας τόνισαν. Φυσικά ο καθένας από εμά είναι σε θέση να υπογραμμίσει κάποιες στοιχές αυτή τη στιγμή. Εγώ όσον με αφορά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως εξάλλου το δείχνουν και πολλές από τις παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι τώρα, είναι το θέμα των της προστασίας των ανηλίκων. Υπάρχουν δύο στοιχεία που πιστεύω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, όχι γιατί δεν υπάρχουν ή δεν αναφέρονται ή τα έχουμε ξεχάσει, αλλά για να ε, πλαισιώσουμε κάποιες στοιχεία. Τα κράτη-μέλη εγγυώνται, λέγεται, σε σχέση με τους ανηλίκους, ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης και πλατφόρμων ε, video sharing θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί το θυμίζω αυτό. Γιατί εδώ σημαίνει συμμετοχή και άμεση ευθύνη των κρατών μελών.

αυτή η διάταξη και ως προς αυτό πιστεύω πως η αναφορά όπως διαρκώς γίνεται στο βλαβερό ε, περιεχόμενο, στη δωρεάν βία, στην πορνογραφία που μάλιστα περιλαμβάνονται από τους ε, ε, σταθμούς και τους παρόχους τηλεοπτικών εκπομπών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η ιδέα του να το ξεπεράσουμε και αυτό είναι, με βρίσκει σύμφωνο και το λέω αυτό και για κάποιες Πιστεύω πως κάποιες παρεμβάσεις υπογράμμισαν την ανάγκη που να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, όσον αφορά τον υποδάβληση μίσους. Εδώ θα ήθελα να πω και εγώ υποβάλλω και εγώ κάποιες προτάσεις, ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να διευκρινίσουμε εδώ το γεγονό ότι υπάρχει μια ολόκληρη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία έκφραση και ενημέρωση που αφορά την υποδάβληση μίσου. Και επί τη βάση του κειμένου τη Επιτροπή, που εδώ είναι ένα εκτιμώντα, ωστόσο εγώ υπογραμμίζω τη συγκεκριμένη αναφορά γιατί έχουμε ήδη κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα μπορούσε να συμπληρώσει αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εξίσου σημαντικό νομίζω πως είναι να θυμίσουμε σε σχέση με το κείμενο της Επιτροπής το γεγονός ότι υπάρχει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαιώματα των ανηλίκων και διαβάζω στο, στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που χρησιμεύουν ως βάση για κάθε νομοθεσία ευρωπαϊκή που αφορά τους ανηλίκους. Υπάρχουν τα άρθρα 5 και 19 της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που ε, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την προστασία των παιδιών σε σχέση με τα οπτικοακουστικά μέσα. Και αυτό βοηθά προς την κατεύθυνση της σύνθεσης που θα κληθείτε να κάνετε με βάση τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ε, περαιτέρω στοιχείο και το διαβάζω γρήγορα ε, αναφέρομαι στις εμπορικέ ε, ανακοινώσεις και εδώ τα κρατη πρέπει ε, να, εξασφαλίσουν και μάλιστα η τροπολογία των δύο συνηγητριών όπως και ε, τα όσα ανέφερα για τις υπηρεσίες που αναφέρουν που αφορούν μάλλον τους ανηλίκους. Ε, υπάρχουν ήδη και εδώ νομίζω πως μια επίσημη πενθύμηση και βεβαίως η οδηγία δεν μπορεί να μην το αναφέρει αυτό, να αποφευχθεί η προσβολή ε, θρησκευτικών ομάδων, μελών, ε, διαφόρων οργανώσεων ή μορφές σεξουαλ, σεξουαλικότητας των παιδιών ή τρόποι υποβάθμισης των γυναικών. Επίσης, το θέμα της πορνογραφίας Όλα αυτά πιστεύω πως εδώ θα πρέπει να αναφερθούν. Αυτά για τις πιο εμπορικές επιτυχίες και για το ηλεκτρονικό εμπόριο να σας πω ότι ναι υπάρχει εκείνη η άλλη οδηγία αλλά όταν συντάχθηκε εκείνη η οδηγία και επειδή είμαστε στον πρώτο γύρο υπήρξε κάποιος που ζήτησε την ενσωμάτωση γνωμοδοτήσεων άλλων επιτροπών σε σχέση με ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί. Γιατί ίσως κάποια πράγματα δεν έχουν ενταχθεί εδώ. Ε, δεν θα ήθελα λοιπόν να λόγω της ύπαρξης κάποιες άλλες οδηγίες να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που ωστόσο τίθενται. Ευχαριστούμε κύριε Μόργαν και εγώ θέλω να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, αλλά Α, ναι, συγγνώμη, ο συνάδελφος Σδροβιεύσκη, με συγχωρείτε. Ναι, ζητήσατε το λόγο προηγουμένω. μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπει ο συνάδελφος να αναφερθώ σε κάτι που δεν συζητηθήκε παρόλο που συζητήσαμε σημαντικά πράγματα. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην εισηγήτρια. Επειδή έχουμε μια τροπολογία εδώ στην έκθεση που αφορά αυτό ακριβώς το σημείο. Βλέπουμε ότι σε διάφορες μάλιστα τροπολογίες υπάρχει με υποχώρηση όσον αφορά τη θέση της έργα και μια ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου. Αυτό μου φαίνεται κάπως αντιφατικό. Ο συνάδελφος Βέντα ήδη μίλησε για την ακύρωση κάποιων τροπολογιών, αλλά να ρωτήσω εγώ το εξής βασικό ερώτημα. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή γιατί ακολουθήσατε αυτή την κατεύθυνση δηλαδή, γιατί το έργο ας πούμε δεν θα έχει πια κάποιες αρμοδιότητες ενώ αντίθετα η Επιτροπή ενισχύεται. Ποια είναι τα επιχειρήματα που σας έπεισαν για να ακολουθήσετε αυτό το, αυτή την κατεύθυνση και να κάνετε αυτή την αλλαγή. Μπορείτε να μου πείτε. Πρόεδρος, θα απαντήσουμε βέβαια μετά οι συγκίτρες. Να πω και εγώ δύο πράγματα ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί νομίζω ότι συζητήσαμε πράγματα σημαντικά. Αφερθήκαμε στις τροπολογίες, στα ανοίγματα, στις συγκλήσεις και να πω ότι νομίζω εγώ ότι είναι σημαντικό το θέμα που αφορά το άνοιγμα για το ζήτημα της διαφήμισης και τους παραγωγούς εκπομπών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει εδώ μια ισοτιμία και μια ισορροπία. Διατηρώντας όμως κάποια όρια σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή και την ποιότητα των έργων, κάτι το οποίο δεν αναφέρουμε συχνά και είναι σημαντικό. Το άνοιγμα δηλαδή που είδα και η αναζήτηση ισορροπίας, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη τους είναι θετικό, αλλά έχουμε υπόψη μας μάλλον ότι υπάρχει μετά και ο έλεγχος αυτών των νέων αντικειμένων που βγαίνουν στο ίντερνετ. Υπάρχουν λοιπόν ανάγκες και θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, να αντέξει το όλο σύστημα όσον αφορά και τα παρουσιακά αλλά και τα νέα μέσα σχετικά με την διαφήμιση ώστε να υπάρχει δηλαδή γενικότερα ισορροπία. Αναρωτιέμαι αν σε σχέση με τις σημαντικές προτάσεις για το φάσμα 8-11, αν εδώ θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι γίνεται, αν τηρείται πραγματικά δηλαδή αυτό το όριο που αφορά αυτό το χρονικό διάστημα. Άλλο ένα ζήτημα αφορά αυτό που έσαι και συνάδελφος Τρούπελ και που νομίζω διευκρινίστηκε Προηγουμένω από διάφορου συναδέλφου και από τις ηγετρίες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Γιατί ακούσαμε και μια ερώτηση εδώ σχετικά. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια ανοίγματα σε σχέση με την ευθύνη για το περιεχόμενο όσον αφορά αυτέ τις πλατφόρμες που ανεβαίνουν τα βίντεο. Δηλαδή ώστε να μην φιλοξενούν μόνο παθητικά αυτά τα βίντεο, αλλά να υπάρχει μια προεπιλογή του περιεχομένου με την συνάδελφο Μόργαν κάναμε μια τροπολογία εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό σημείο γιατί θεωρώ ότι αποτελεί ακριβώς αυτό το λεπτό ζήτημα που αφορά ευθύνες οι οποίες δεν πρέπει να επαφείται μόνο σε παθητικούς αλγόριθμους αλλά στην ενεργό επιλογή του περιεχόμενου. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν, γι' αυτό το σημείο θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις εγώ ώστε να υπάρχει έτσι μια ισορροπία. Τρίτο σημείο και σταματώ. Το θέμα των ανηλίκων. Εγώ κατέθεσα προσωπικά τροπολογίες ιδιαίτερα από αυτήν την οριζόντια ομάδα για τους ανήλικους θα έλεγα να αφήσουμε την απαγόρευση όσο έχει αυτή τη στιγμή στην οδηγία γιατί είναι σημαντική που αφορά ακριβώς τις εκπομπές και τους ανήλικους Και αυτό επειδή κυρίως όλες οι χώρες μέλη έχουν ερμηνεύσει πολύ αυστηρά, όσο πιο αυστηρά γίνεται, την τρέχουσα οδηγία. Αντίθετα λοιπόν με αυτό που υπόθηκε κάπου, το θέμα όμως που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να προβλέψουμε, και αυτό ακριβώς προτείνουμε, να προβλέπουμε όχι μόνο να έχουμε κάποιες μορφές προστασίας χωρίς μετά να ευκρινίσουμε το πώς θα εφαρμόζονται αλλά να αφήνουμε τις εθνικές αρχές να καθορίζουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι κώδικοι της οδηγίας εφαρμόζονται και υπάρχουν και κυρώσεις. Αλλιώς θα συζητάμε για κάτι το οποίο είναι γενικόλογο και αόριστο. Μετά, για τις αρχές και την έργα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα εδώ από τις εισηγήτρες δηλαδή. Ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο ότι αυτά τα δύο αντικείμενα έργα και ρυθμιστικές αρχές είναι συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής όχι μόνο το ένα έτσι και αυτό το διευκρινίζω ότι υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις και για τις αρχές χαίρομαι που υπήρξε έτσι, ένα βήμα πρόοδου εκ μέρους όλων σχετικά με το γεγονό ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει στην πράξη και λειτουργικά αλλά και νομικά πρέπει να είναι ανεξάρτητες. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στις διάφορες χώρες. Δεν το αφισβητεί κανεί αυτό. Η γενική όμως αρχή πρέπει να είναι σαφής. Αν υπάρχει βοήθεια από τις κυβερνήσεις και τι χώρε, πολύ ωραία. Αλλά πρέπει για αυτό το σημείο να υπάρχει ένα σωστό άνοιγμα και μια διευκρίνηση. Και νομίζω είναι καλό να γίνει αυτό γιατί μας ενδιαφέρει όλους αυτό το σημείο και θα ήταν καλό να δούμε ποιες θα ήταν οι πιθανές διέξοδοι για την ανέβρεση λύση εδώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο Αλότσο από την Επιτροπή και να την ευχαριστήσω που ήρθε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Για τι πλατφόρμε ανταλλαγή βίντεο καταρχά. Υπάρχει μεγάλη παρανόηση εδώ και πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν μιλάμε για αυτές τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, λέτε ότι πρέπει να γίνεται προεπιλογή του περιεχομένου πριν να ανεβεί αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για μια υπηρεσία με άλλες δυνατότητες, δηλαδή ένα κανάλι του YouTube το YouTube ας πούμε το οποίο έχει δικιά του υπηρεσία για τα παιδιά και τα λοιπά και κάνει δικό του έλεγχο και τα λοιπά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η έλεγχη είναι η έλεγχη του video on demand. Όταν μιλάμε για αυτές τις πλατφόρμες, την πρόταση της Κομισιόν αυτές, μιλάμε για πλατφόρμες που δεν κάνουν εκ των προτέρων έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο που ανεβαίνει. το περιεχόμενο προέρχεται από τους χρήστες. Μπορεί να πούμε το βίντεο των γενεθλίων του Γιώκα Και να ζητήσουμε λοιπόν από μια πλατφόρμα ανταλλαγή βίντεο εκ των προτέρων να ελέγξουν αυτές 400 ώρες ένα λεπτό που ανεβαίνουν καθημερινά μου φαίνεται αδυνατό. Δεν γίνεται τεχνικά να εφαρμοστεί αυτό και δεν θα εφαρμοστεί. Είναι αδύνατο να το λέξει η πλατφόρμα και είναι αδύνατο ο ρυθμιστή να το εφαρμόσει αυτό. Οι ρυθμιστέ, ήδη σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρέ ε, δυσκολίε για την εφαρμογή αυτών των κανόνων για το video on demand. Φανταστείτε τώρα να πάμε σε τέτοιες καταστάσει. Εντάξει, να έχουμε την παρά γιατί διατηρώντας αυτά προβλέπει η οδηγία για τις πλατφόρμες τις εμπορικές κτλ. Αλλά ε, φανταστείτε μετά να το επεκτείνουμε και να πούμε ε, για το περιεχόμενο αυτού του είδους με το βίντεο του Γιώκα μου κατά το, το οποίο θα πρέπει να λέγεται κατά πόσο περιέχει βία κλπ. κλπ. Δηλαδή ζητάμε στην ουσία να κάνουν ένα προέλεγχο οι πλατφόρμες. Το γεγονό λοιπόν ότι η Κομισιόν ζητά έλεγχο συμβατότητας δίνει ότι θεωρείται έχει αποκλειστικά δίκιο, αλλά επειδή θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί εκεί. Το ίδιο και με τους κανόνες της διαφήμισης. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρχει αναγγελέχου του, της διαφήμισης στο YouTube, αλλά ίσως όχι όταν έχουμε να κάνουμε χορηγία ή με τοποθέτηση προϊόντων, γιατί για τους δημιουργούς αυτών εκπομπών ίσως να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεση σε περίπτωση που δεν έχουν παράξει ήδη αυτή την εκπομπή. Φανταστείτε λοιπόν όταν έχουμε να κάνουμε κάποιον ο οποίο δεν έχει έλεγχο πάνω σε ένα προϊόν και ο οποίο ε, αποφασίζει να μην ισχύουν κάποια πράγματα για τους παραγωγούς αυτού του περιεχομένου. Οπότε εμείς εδώ θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μα, να έχουμε σωστού στόχου, να προστατεύσουμε του καταναλωτέ μα αλλά οι τεχνικές πτυχές να τις έχουμε κατά νου γιατί οι κανόνες πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζονται. Με καθησυχάζει αυτό που άκουσα για την εξαρτησία των ρυθμιστών για τη σημασία των κανόνων εδώ για τη σημασία ας πούμε του να υπάρχουν ρυθμιστές οι οποίοι είναι νομικά μακριά ή χωριστά από τις κυβερνήσεις το ίδιο και για την έργα ότι πρέπει να είναι κάτι το τελείως χωριστό από τι υπόλοιπε μονάδε εμπειρογνωμών και μην υπόκειται σε κανένα πολιτικό έλεγχο. Αυτά είναι θετικά. Για τη διαφήμιση είναι αλήθεια ότι η εντολή για την Κομισιόν στα πλαίσια του Ρεφιτ ήταν το να δούμε κατά πόσο υπάρχει εδώ δυνατότητα ευελιξία. Αυτό λέμε εδώ πέρα. Αν δεν υπάρχει ευελιξία θα έχουμε περισσότερο κανονιστικό πλαίσιο παντού. Πάντως να θυμάστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια οδηγία ελάχιστη εναρμόνιση. Δηλαδή, αν η εξέλιξη στην αγορά που βλέπουμε, η οποία σημαίνει ότι αυτοί που παράγουν αυτά τα μέσα αυτορυθμίζονται. Γιατί αν υπάρχει πολλή διαφήμιση θα φύγει ο κόσμο και θα αρχίσει να βλέπει Netflix που δεν έχει διαφήμιση. Θεωρούμε λοιπόν ότι στις ε, χώρες με ακόμα δεν έχει ε, εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση αγορά, οπότε μπορούν να επιβληθούν αυστηροί οι κανόνες. Αλλά δεν υπάρχει ένα ελάχιστο, τότε δεν θα είναι δυνατό να γίνει αυτό σε αγορές όπου ε, έχει υπάρξει μεγαλύτερη εξέλιξη. Και να θυμάστε ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης περιεχομένου είναι η διαφήμιση. Τώρα για την πρόθεση των ευρωπαϊκών έργων. Δασμοί. Να διευκρινίσω ότι εδώ απλά και μόνο διευκρινίζουμε αυτό που λέει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Η νομοθεσία που ισχύει. Και λέει ότι αυτό το είδο τέλο πάντων περιορισμών και θα το δείτε αυτό σε διάφορες ε, αποφάσεις της ε, Κομισιόν που αφορούν εθνικές καταστάσεις εκεί έχει διευκρινιστεί ότι αυτό τέλο πάντων δεν είναι υποχρεωτικό απλά και μόνο αποτελεί μια δυνατότητα για τις χώρες μέλη. Ένα άλλο δηλαδή είδος εισόδων για τη χρηματοδότηση του περιεχομένου αυτή η δασμή. Θα μπορούσα να πω και παραπάνω, αλλά δεν θέλω να σας φάω χρόνο. Διαδικασία εξαιρέσεων. Γιατί είδα κάποιες ιδέες που λένε, ας πούμε, μία παράβαση και μόνο να επιθυμίσουμε ότι αν ζητήσουμε στην οδηγία επαναλαμβανόμενε ε, παραβάσεις, τρεις ας πούμε, τότε εδώ έχουμε μια παρέκκληση στις βασικές ελευθερίες και το να αναστείλουμε τη λειτουργία ενό καναλιού που λειτουργεί διασυνοριακά μου φαίνεται πολύ ακραίο λύση. Γι' αυτό ακριβώ την πρόταση, ω έχει σήμερα, ζητάμε να υπάρχουν τρει παραβάσει αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη, όπου υπάρχει κάτι το έκτακτο και μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πιο ταχεία διαδικασία. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ ειλικρινά δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι χαμένη αυτή η ευκαιρία, ακόμα και για την υπόδειξη ευθυνών. Το λέγαμε πριν. Ακόμα και αν κανεί δεν θέλει να θέσει δυσκολίε στι πλατφόρμες, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είναι ουδέτερα σύνολα περιεχομένου, αλλά πραγματικοί ανταγωνιστέ στην αγορά. Και αυτό είναι ο κίνδυνο να χάσουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερα ισότιμο πεδίο. Level playing field. Αυτά ήθελα να πω και τώρα η συγγήτρης ποια θα πάρει πρώτη το λόγο. Η Σαμπίνα. Ναι, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και των άλλων πολιτικών ομάδων για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα για το πώς έχουν οι θέσεις του καθενός που μεταβάλλονται και αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πράγματα που είπαμε και την τελευταία φορά ως εισηγήτριες στην περασμένη συνεδρίαση. Έχουν προκύψει νέα δεδομένα, νέες εξελίξεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποδυνάμωση του έργα και την ενίσχυση ε, της λεγόμενης ε, πολιτική ε, επιτροπή επαφής που είπε και ο κύριος Κρασνοντέψκη. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να αποδυναμώσουμε την έργα, αλλά να βρεθεί η χρυσή τομή και η ισορροπία ανάμεσα στα τεχνικά ζητήματα και τις ανταλλαγές και τη ρυθμιστική αρμοδιότητα που έχει η έργα. γιατί διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα και είπαμε ότι υπάρχει η ομάδα επαφής αλλά και οι έργα που θα πρέπει να ε, συνεννοούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να περνάνε ακρόαση και τα λοιπά. Εξού και η τροπολογία 82 και έτσι θα πρέπει να την αναλυφθούμε, όπου τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρύτατη πολιτική αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σε εθνικό κρατικό επίπεδο δηλαδή. Να γνωμοδοτεί η Επιτροπή Επαφής. Και από την άλλη και η έργα θα πρέπει να γνωμοδοτεί, το είχαμε πει από την περασμένη φορά. Μας είχε διαφύγει, ήταν λάθο. Η έκθεση έργα βεβαίως δεν θα πρέπει να καθορίζεται από την ομάδα επαφής, Θα πρέπει να συνεννοούνται και να λαμβάνουν γνώση οι επιτροπές ε, των εκθέσεων για να έχουν όλη την ίδια πληροφόρηση. Αυτό ήταν ένα λάθος που κάναμε, αλλά θα τη διορθώσουμε με τροπολογίες. Ερωτήσατε όμως, αν κατάλαβα καλά, κάτι για την τροπολογία 85, όπου είπαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν ε, άποψη για το περιεχόμενο, για ε, τη συντακτική, την εκδοτική γραμμή κτλ. Αυτό είναι σωστό. Ε, αρμόδια ρυθμιστική αρχή δεν ελέγχει τι θα γράφεις και πώς θα έχει σύνταξη της είδηση ή του περιεχομένου, αλλά εάν το πρόγραμμα που εκπέμπεις ανταποκρίνεται στις ε, προϋποθέσεις που έχεις βάλει. Εδώ μιλάμε για ελευθερία του τύπου και ελευθερία των δημοσιογράφων. Δεν θα του πεις εσύ τι θα εκπέμπει και ελευθεροτυπία λοιπόν και ελευθερία στην έκφραση. Αυτό που κάνει η ρυθμιστική αρχή είναι ελέγχει εάν τηρούνται οι ε, υποχρεώσεις με βάση τον νόμο. Αλλά ούτε η εκδοτική γραμμή, ούτε ο συντακτικός, ε, στα συντακτικά της ε, κάθε εκπομπής. Δεύτερο σημείο αξιολόγηση εξάντα ή εξπόστ, εκ των προτέρων εκ των υστέρων και σε πλατφόρμες video sharing. Το ίδιο ισχύει αυτό. Δεν πρόκειται για εκ των προτέρων έλεγχο ε, ενός βίντεο. Δεν θα πρέπει η πλατφόρμα να κοιτάξει τι επιτρέπεται να εκπέμψω ή όχι, αλλά εκ των υστέρων να υπάρχει δυνατότητα ε, ότι, να λέμε ότι αυτό βλάπτει τους νέους ή μπορεί να είναι απειλή για τους ε, ανηλίκους. Οπότε να το ε, προβάλλεται μια ώρα που υποτίθεται ότι δεν βλέπουν ανήλικοι. Υπάρχουν κώδικες δεοντολογίας στην αυτορύθμιση που θα πρέπει να τηρούνται και σε πλατφόρμες video sharing για να παραμένει η προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών γενικότερα εξασφαλισμένη. Αλλά αυτά είναι εκ των υστέρων, όχι εκ των προτέρων όπως και στα τηλεοπτικά προγράμματα, δεν είναι ποτέ εξάντα, είναι πάντα ex post. Κανονικά δεν μπορεί να υπάρχει προληπτική ε, παρακολούθηση και έλεγχος για να δω τι πρόγραμμα έχει, όχι αυτό δεν θα το εκπέμψεις, αλλά αυτή τη στιγμή σε εκπαιμφθεί να τραβάει και καν αυτή η Επιτροπή. Και κατά τα άλλα με χαρά θα παρακολουθήσω και τις συζητήσεις και ε, θα συνεργαστώ με τους ε, σκιώδης Είμαι αισιόδοξη ότι θα καταλήξουμε και μάλιστα ομόφωνα. Ε, η Πέτρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ε, και τους και ηγητές μας, αλλά και όλους τους άλλους που μίλησαν. Ήταν καλή συζήτηση. Κρίμα που έχουν φύγει μερικοί σκιώδεις τώρα. Θα ήθελα να τονίσω κάτι να τα πείτε και στον κύριο Ρούα και στην κύριο Τούν. Κανείς δεν θέλει λογοκρισία εκ των προτέρων έλεγχο. Προς Θεού. Όποιος με ξέρει ε, θα σας πει ότι έχω αλλεργία σε οτιδήποτε μυρίζει λογοκρισία, όχι να συμβαίνει κιόλας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πούμε πραγματικά το εξής. Όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα περιεχόμενο παράνομο, υποδάβληση μίσους, ε, επικίνδυνο ε, ή που παραβιάζει ε, τους κανόνες για τη διαφήμιση, εφόσον το μάθει ο πάροχος θα πρέπει να δράσει. Αλλά μόνο εκ των υστέρων. Είναι σωστό αυτό που λες Χέλγκερ Από ποια στιγμή και μετά, δηλαδή από τον αλγόριθμο, ήδη ένας αλγόριθμος που δεν είναι προϊόν αναζήτησης. Αλλά κάποιος έχει ανεβάσει ένα περιεχόμενο ε, με μορφή διαφήμισης για να κερδίσει χρήματα. Από ποια στιγμή θεωρείς ότι ο πάροχος έχει λάβει γνώση. Αυτό είναι ένα καθόδες ερώτημα. Και αυτό με ενδιαφέρει και εμένα. Να πω ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει λάβει γνώση ο πάροχος και μπορεί να απαιτήσει κανείς να αντιδράσει. και πώς θα βρεθεί αυτή η λύση και η ρύθμιση για να αποδείξουμε ότι ήταν σε γνωστού. Γιατί και οι πλατφόρμες για το video sharing, video on demand ή κλασική επιγραμμική τηλεόραση δεν παίρνουν πάντα στον κορσέ τη διαφήμιση. Βεβαίω η διαφήμιση θα πρέπει να είναι ξεχωριστή και διακριτή και να ξέρει ο καθή ε, ότι άλλο είναι η είδηση και άλλο είναι η διαφήμιση. Και να το... Αυτό είναι λογικό και δεν είναι και ανάρμοστο να το απαιτήσουμε ούτε υπερβολικό. Το ίδιο ισχύει και για τα, τους λόγους μίσους και ε, για τους ανήλικους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ένας από τους λόγους ε, που ε, έβαλε η Κομισιόν στην οδηγία αυτή και το video sharing. Θα βρούμε κάποιο τρόπο για την ευθύνη. Και εγώ με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης δυσκολεύομαι να βάλω και το facebook. Να το ξανασυζητήσουμε με όλους εκείνους που το πρότειναν. Προς το παρόν δεν έχω πιστεί ότι είναι καλή ιδέα ούτε για τον τζόγο. Είμαι πεπισμένη. Θέλει προσοχή αυτό. Θέλετε τόσο να ξεχυλώσουμε τον ορισμό της οδηγίας και το πεδίο εφαρμογής να είναι αρμόδια για όλα και για τίποτα και να μην ξέρει κανείς το λόγο ύπαρξής της. Για την ομάδα έργα ναι, καθεν λέμε εμείς ε, ότι θέλουμε ανεξαρτησία των ε, ρυθμιστικών αρχών. Είναι πάρα πολύ σημαντική αξιολογούμε και τιμούμε και τη δουλειά που κάνει η έργα και στη συγκεκριμένη οδηγία να τα κωδικοποιήσει αυτά. Αυτό τον καιρό λειτουργεί σε ένα νομοθετικό κενό. Θα πρέπει να της δώσουμε μια νομική βάση για να λειτουργεί σωστά. Μπορεί κάπου να υπερβάλαμε, μπορεί να έχουμε κάνει και λάθη. Με τώρα και με δικές μας τροπολογίες θα έχουμε διορθώσει αυτά που Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο. Για τη διαφήμιση θα προσπαθήσω και πάλι να σας πω για την ελαστικοποίηση. Δεν υπάρχει τομέας που να ρυθμίζεται τόσο πολύ όσο ε, τα online για τη διαφήμιση. Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας μπορεί να κάνει ε, όση διαφήμιση θέλει μπορεί να διακόπτει περιεχόμενο, μπορεί να πετάγεται ένα παράθυρο με διαφήμιση κτλ. Όλα επιτρέπονται. Είναι δυνατά. Αν όμως ένα ιδιωτικό κανόν, ε, κανάλι κάνει διαφήμιση, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα όταν έχει καλό περιεχόμενο να βγάζει λεφτά και από τη διαφήμιση, γιατί από εκεί βγαίνει. Δεν μπορεί ο ένας τομέας να έχει υπερβολικά δρακόντιες ρυθμίσεις και ε, νομοθεσία και ο άλλος να είναι τελείως ασίδωτος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είτε θα υπάρχει ποθενά ρύθμιση ή θα υπάρχει αυστηρή και στα δύο. Εμείς δεν θέλουμε να είναι όλα ασίδωτα. Άρα, στην επιγραμμική τηλεόραση τουλάχιστον να υπάρξει μια στοιχειώδης ευελιξία. Δεν είναι και αυτό τίποτα απρεπές. Δεν διευρύνουμε ούτε αυξάνουμε ε, το χρόνο της ε, διαφήμισης. Ίσως καλύτερα είναι να, να έχεις ένα διαφημιστικό σποτ ε, κατά τη διάρκεια μιας ταινία παρά δεκάλεπτη διακοπή για διαφήμιση. Είναι και προς το συμφέρον του καταναλωτή αυτό και του τηλεθεατή. Και ακόμα και τα 30 λεπτά θέλετε να το σκεφτούμε. Αλλά να πεμπολίσουμε τελείως τις υποσχέσεις μας και τις επιθυμίες μας που είπαμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν το βλέπω σωστό. Πώς να το πω. Θα ήταν λίγο ανάρμοστο και αναξιοπρεπές. Το έχουμε πει επανειλημμένα και όχι μόνο προηγούμενη θητεία και η τωρινή με μεγάλη πλειοψηφία. Πρέπει να βρούμε έναν δρόμο. Την αρχή την έχουμε κάνει. Να μην γίνονται όλα στα prime time, σε χρόνο υψηλής τηλεθέασης, ε, να βάλουμε αυτή τη ρύθμιση για να υπάρχει ελεύθερη δυνατότητα κατανομής. Καλά, μισή ώρα συνεχόμενη διαφήμιση δεν υπάρχει κανάλι που να τη βάζει γιατί ε, ξέρουν ότι θα κάνει ο κόσμος ζάπινγκ. Δεν θα κάτσει κανείς να βλέπει μισή ώρα διαφημίσεις. λέει κάποιος ε, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον διθελατή να ε, μην βλέπει τις διαφημίσεις. Μπορεί να το κάνει και τώρα, να αλλάξει κανένα άλλη. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε κάπου και να έχουμε μια καλή οδηγία και να κρατήσει τουλάχιστον καμιά δεκαετία, να μην τα ξυλώνουμε κάθε τρεις και λίγο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις δύο Εμένα μου άρεσε πολύ η απόψινη συζήτηση και το κλίμα που επικράτησε. Χρειαζόταν η απόψινη συνάντηση, ήταν χρήσιμη. Και σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ την Επιτροπή που παρακολουθεί από κοντά αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση και σας λέω ότι η επόμενη μας ε, συναδρίαση προβλέπεται στις 28 Νευρίου στις 3. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς. Ε, γεια σας.